Συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Έχουμε δύο σημεία στην μερίσια διάταξη πριν ε, περάσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών. Πρώτον, παρουσίαση μελέτης για τα χρηματοδοτικά μέσα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, όπου έχουμε τον κύριο Χάιμφαν Έσεν εδώ πέρα από το Delft και τον κύριο Ρόμπερτ Μπέιν από την ITS στο Leeds. Το Leeds είναι στην άλλη μεριά των βουνών εκεί πέρα από τα δικά μου τα πατρογονικά και θα μας παρουσιάσουμε εδώ πέρα τα σχετικά. Σας παρακαλώ λοιπόν γύρω στα 10 λεπτά για να ε, κάνουν και ερωτήσεις οι βουλευτές. Ποιος θα ξεκινήσει. Α, μία, μία παρουσίαση θα γίνει. Μάλιστα. Ε, τότε έχετε 20 λεπτά. Ωραία. Παρουσίαση της μελέτης για τα χρηματοδοτικά μέσα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Κύριε να έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας καλέσατε να σας κάνουμε αυτή την παρουσίαση για τα χρηματοδοτικά μέσα. Κάναμε μια μελέτη την CE Delft με την ITS Leeds και σε συνεργασία με την ε, TPR e ένα, μια άλλη οργάνωση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Βασικός στόχος της μελέτης αυτής ήταν ε, να δώσουμε μια γενική εικόνα των χρηματοδοτικών μέσων και των πηγών χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή υποδομή μεταφορών, ειδικά αναφερόμενη στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Σε τελική ανάλυση οι υποδομές πληρώνονται από τους χρήστες ή τους φορολογούμενους, αλλά κοιτάμε να δούμε εδώ πέρα τις λεπτομέρειες. Κοιτάξαμε και τα σχετικά ζητήματα, την στρατηγική ευθυγράμμιση και την επιχειρησιακή ευθυγράμμιση αυτών των μέσων και ζητήματα που φορούν τη διοικητική ικανότητα. Αξιολογήσαμε επίσης τις διάφορες επιλογές ε, των προσφάτων προτάσεων της ε, Κομισιόν, τις κατευθυντήριες γραμμές ε, και όλες τις υπόλοιπες προτάσεις που βασικά σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των δικτύων αυτών. Και επίσης διατυπώσαμε συστάσεις πολιτικής με βάση την αναλυσή μας και... Three, uh, Είπα, αυτό έγινε από τους τρεις ε, συνεταίρους ε, της κοινοπραξίας μας. Για να ξεκινήσω γρήγορα, η πολιτική αυτή είναι σημείο κλειδί της πολιτικής μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και κάποιες δεκαετίες. Καλό είναι να επιθυμίσουμε τους βασικούς στόχους αυτής της πολιτικής σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, τη βελτιωμένη προσβασιμότητα για επιβάτες ε, και φορτίο και κάτι το οποίο τελευταίως έγινε πιο σημαντικό, στόχοι περιορισμού της κλιματικής ε, αλλαγής. Επίσης, οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, σημαντική στόχη της πολιτικής αυτής και Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως στοχεύει ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δηλαδή δίκτυα τα οποία έχουν προστιθέμενη αξία για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ορισμός των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών είναι όλε, όλες οι υποδομές που εξυπηρετούν τις μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών και η πολιτική μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει συνεισφορές της Ένωσης και στην ε, ε, τωρινή χρηματοδοτική περίοδο μιλάμε για 52 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα σοβαρό ποσό ε, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οπότε εδώ πέρα έχουμε μία παρουσίαση του κόστους και της χρηματοδότησης των ε, δικτύων αυτών στην τωρινή χρηματοδοτική περίοδο, την προηγούμενη και την επόμενη και βλέπετε πως οι αριθμοί αυξάνονται. Τα 52 που ανέφερα είναι στη δεύτερη στήλη, το σύνολο των ε, κονδυλίων, ε, δύο ευρωπαϊκών δικτύων συνοχής και ΕΤΠΑ, έχουμε δηλαδή την άμεση χρηματοδότηση της Ένωσης, Υπάρχει, υπάρχουν και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που συνολικά ήταν 41 δισεκατομμύρια στην περίοδο 2000-2006 και έφτασαν τα 53 ε, τελευταία εκτίμηση που βρήκαμε. Στην τωρινή περίοδο χρηματοδότησης βλέπετε επίσης στην κορφή πως το συνολικό κόστος, η συνολική χρηματοδότηση αυξάνεται από 300 δισεκατομμύρια το, στην περίοδο 2000-2006 σε 390 στην τρέχουσα περίοδο και υπολογίζεται πως θα φτάσουν τα 540 δισεκατομμύρια στην επόμενη χρηματοδοτική περίοδο για να επιτύχουμε τους στόχους. Σημαντική αύξηση. Επίσης λέμε πως ε, είναι η κατανομή μεταξύ των 15 της Ένωσης και των 12 νέων μελών και βλέπετε πως ένα σημαντικό μέρος ε, εξοδεύεται στα παλαιά κράτη-μέλη ε, και τα δύο αυξάνονται ούτως ή άλλως. Τώρα εδώ κάποιες πιο λεπτομερείς ε, πληροφορίες μπορείτε να τις δείτε στην έκθεση για τα διάφορα μέσα. Βλέπετε πως το ίδιο το πρόγραμμα αριθμεί 8 δισεκατομμύρια είναι πολύ μικρότερο από το ποσό που είναι διαθέσιμο από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής. Αυτά τα δύο μαζί είναι πάνω από 80 δις και συμπεριλαμβάνει βεβαίως και κάποιες άλλες υποδομές μεταφορών. Βλέπετε το τι είναι ε, διαθέσιμο. Μιλάμε για γύρω στα 44 δισεκατομμύρια. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, δίνει περισσότερα, γύρω στα 53 δισεκατομμύρια και βλέπετε πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Αυτές είναι, αυτό είναι το μέγιστο ποσοστό, π.χ. Ε, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών μιλάμε σε κάποιες περιπτώσεις για μελέτες. Στις άλλες περιπτώσεις είναι χαμηλότερο το ποσοστό συγχρηματοδότησης εδώ πέρα βλέπετε κάποιες πληροφορίες, το τι καλύπτεται από τα κράτη-μέλη. Στα αριστερά βλέπετε πως από τα 390 δισεκατομμύρια σε αυτή την περίοδο χρηματοδότησης τα 3 τέταρτα καλύπτονται από άλλες πηγές που συμπεριλαμβάνει και επενδύσεις από επενδυτές εθνικές κυβερνήσεις και περιφερειακές κυβερνήσεις. Από το υπόλοιπο τέταρτο, 14% είναι Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το υπόλοιπο είναι Ταμείο Συνοχής, ΕΤΠΑ και Διευρωπαϊκά Δικτύα Μεταφόρων. Στα δεξιά βλέπετε την κατανομή μεταξύ των προτεραιοτήτων, των έργων προτεραιοτήτων και των λοιπών έργων και βλέπετε πως ε, το πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών εστιάζεται σε έργα προτεραιοτήτων ενώ στα υπόλοιπα η κατανομή είναι διαφορετική μεταξύ προτεραιοτήτων και μη. Εδώ πέρα έχουμε μία παρουσίαση του τι ξοδεύεται στα βασικά, στους βασικούς, στα βασικά μέσα Βλέπετε εδώ πέρα πως το ποσό που ξοδεύεται στους σιδηρόδρομους και τους δρόμους είναι ίδιας τάξης μεγέθους. Πολύ λιγότερα σε ε, διατροπική μεταφορά και σε πλεύσιμους ποταμούς. Επίσης ενδιαφέρον είναι το ότι η μερίδα του Λέοντος πηγαίνει στους σιδηρόδρομους, ενώ στο Ταμείο Συνοχής ε, το ποσοστό των οδικών μεταφορών είναι πολύ ψηλότερο. Εδώ πέρα έχουμε πολύ πιο λεπτομερή δεδομένα. για το ΕΚΠΑ και το Ταμείο Συνοχής ε, από το 2007 μέχρι το Σεπτέμβριο 2010 βλέπετε πως υπάρχουν και κάποιες διαφορές στο τι έχει εγκριθεί και το τι έχει ήδη κατανεμηθεί σε συγκεκριμένα έργα. Ένα μέρος έχει ήδη πάει σε συγκεκριμένα έργα για αυτοκινητόδρομους ε, και για εθνικούς νόμους είναι κατά τη ψηλότερο από ό,τι για τους σιδηρόδρομους. Να σας δώσω μια ιδέα τώρα του πώς λειτουργεί για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων. Πήραμε το έργο προτεραιότητας υπαριθμών 6 Σιδηρόδρομος από την του στο Μπορντό στη Γαλλία, συνολικό ποσό 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Βλέπετε εδώ πέρα πως υπάρχουν διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης από την RFF, το Γαλλικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, το Γαλλικό Δημόσιο, 3 δισεκατομμύρια, ε, οι μέτοχοι εμπορικές τράπεζες, 1,6 δις, με εγγύσει του γαλλικού δημοσίου, βλέπετε πως είναι πολύπλοκη η χρηματοδότηση και χρησιμοποιούνται πολλά και διάφορα μέσα σε αυτές τις ε, περιπτώσεις. Για την επόμενη λοιπόν χρηματοδοτική περίοδο είχαμε 8 δισεκατομμύρια στο πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, το οποίο θα αντικατασταθεί από το μέσο συνδέοντα την Ευρώπη, στο οποίο η πρόταση κομισίων περιλαμβάνει 31,7 δισεκατομμύρια, ποσό πολύ σημαντικότερο. Οπότε έχουμε άλλα 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής και Αυτό το οποίο υπολογίζουμε εμείς μετά το σύνολο είναι 41 δις, κάτι το οποίο υποθέτει βεβαίως πως το ποσό για τις μεταφορές μέχρι το 2020 θα είναι το ίδιο στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Αν προσθέσουμε λοιπόν τα δύο, μιλάμε για 31 συν 31, γιατί το, το, το 41 είναι, ε, περιλαμβάνει 10 ε, ήδη δις. Οπότε μιλάμε για 63 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια γιατί εξαρτάται από την ζήτηση. Σημαντικό στοιχείο αφορά και τα ομόλογα έργων. Δεν θέλω να μπω τώρα σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά πρέπει να το αναφέρω σύντομα. Το σκεπτικό λοιπόν είναι να βελτιωθεί η φερεγγιότητα των έργων για να προσελκύσουν οι ιδιώτες ε, επενδυτές, να υπάρξουν κάποιες εγγυήσει για να περάσουν κάποιοι κίνδυνοι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με αυτές τις εγγυήσει λοιπόν υπάρχει ένας πολλαπλασιαστής ε, και λένε πως για κάθε δισεκατομμύριο το οποίο ξοδεύεται αναμένεται να προσελκυστεί, να προσελκυστεί ποσό από άλλους επενδυτές ε, σε ποσό 15 πλάσιο και 20 πλάσιο. Οπότε αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Το επιχείρημα λοιπόν εδώ πέρα, όταν σχεδιάζουμε τέτοια μέσα, είναι οπως η αγορά έχει αποτυχίες και δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. Οπότε δεν ε, λάβαμε μία απάντηση για το ποια ακριβώς αποτυχία της αγοράς αντιμετωπίζεται έτσι. Θεωρούμε λοιπόν πως υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα που πρέπει να έχουμε κατά νου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πιλωτική φάση 2013. Ε, μιλάμε για 220 εκατομμύρια που είναι το μάξιμο ποσό το οποίο μπορεί να διατηθεί. Επίσης υπάρχει και το στοιχείο των ΣΔΙΤ όπου κάναμε μια αξιολόγηση του πώς έχει χρησιμοποιηθεί και το ποιες είναι οι εμπειρίες με τα έργα ΑΣΔΙΤ. Ο συναδελφός μου, ο κύριος Μπέιν, είναι από τους ειδικού στον τομέα αυτών και καταλήξαμε στο ότι είναι εποφελής οι δίτα, αλλά μόνο εάν εφαρμοστούν ε, σωστά και με σωστές ε, συμβουλές περί δημοσίων προμηθειών. υπάρχουν και κίνδυνοι, εξαρτάται λίγο από τον τύπο του ΣΔΙΤ που επιλέγετε Ανάλογα λοιπόν με το εάν μιλάμε για πληρωμές ανάλογα με την απόδοση του έργου και βεβαίως δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται τα ΣΔΙΤ για να φεύγουν τα έργα από τους ε, ισολογισμούς των κυβερνήσεων. Τώρα να περάσουμε στις προτάσεις με βάση την ανάλυση που κάναμε τα συμπεράσματα από την εξέταση της πολιτικής η οποία έγινε το 2009-2010 ήταν πως πολλά έργα προτεραιότητας έχουν μείνει πίσω όσον αφορά το πρόγραμμα και ένας λόγος είναι βεβαίως η ανεπαρκής χρηματοδότηση. Επίσης ε, η εξέταση κατέληξε ότι χρειάζεται περισσότερη προσοχή για τις διασυνοριακές διασυνδέσεις. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα είναι, αν θέλετε, έχουν μια μορφή εμβαλωματική ε, εθνικών έργων χωρίς ε, διασύνδεση. Επίσης η διαλειτουργικότητα που είναι ζήτημα ειδικά για τους σιδηρόδρομους και τις διατροπικές μεταφορές. Τώρα, εάν δείτε τις νέες προτάσεις, έχουν αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Συνοψίζοντας, θα λέγαμε τα εξής. Βλέπετε πως ε, αυτά τα διάφορα μπαλώματα τα αντιμετωπίζουμε όχι μόνο ορίζοντας έργα προτεραιότητας, αλλά ένα κύριο δίκτυο, κάτι το οποίο είναι ο βασικός στόχος για να αναπτυχθεί. Οπότε έχουμε μια αρκετά σημαντική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη πολιτική. Άλλο στοιχείο είναι το ότι τα 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής έχει οριστεί να πάνε στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, κάτι το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε πως δίνει ακριβώ μεγαλύτερη προτεραιότητα στο δίκτυο το βασικό. Έχουμε και τα ομόλογα έργων και η πρωτοβουλία αυτή ε, είναι σημαντική για να επενδυθούν χρήματα στα δίκτυα και τέλος η στρατηγική ευθυγράμμιση των διαφόρων ταμείων και έχει συμπεριληφθεί σε προτάσεις. Θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό. Αν δούμε λοιπόν στρατηγική ευθυγράμμιση μπορείτε να δείτε πως οι στόχοι και οι προτεραιότητες των μέσων έχουν ευθυγραμμιστεί πλέον πολύ ε, καλύτερα και μιλάμε για διασυνοριακά έργα, διαλειτουργικότητα και την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Αναφέρονται οι στόχοι επίσης. Βλέπετε πως ε, με την δέσμευση αυτών των 10 δισεκατομμυρίων θα δοθεί περισσότερη προτεραιότητα στα κύρια δίκτυα και έχουμε και υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης 10% περισσότερο για έργα ε, που επηρεάζουν το κλίμα και είναι διασυνοριακά και η πολιτική συνοχής η οποία συμπεριλαμβάνει την αιρεσιμότητα εξ άντε. Βεβαίως, αν δούμε ολόκληρη την πρόταση, αυτό το οποίο λείπει είναι πως ε, δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συνεισφορά των νέων προτάσεων αυτών ε, στη μείωση εκπομπών και στον διαχωρισμό των διαφόρων μέσων μεταφοράς και δεν είναι σαφές προτάσεις. Ένα άλλο θέμα βέβαια είναι και η επιχειρησιακή ευθυγράμμιση. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως ε, η εστίαση σύστημας μεταφοράς ε, αυτή τη στιγμή είναι διαφορετική, το είδατε και πριν, βλέπετε πως το πρόγραμμα ευρωπαϊκών δικτύων περισσότερη χρηματοδότηση πάει στον σιδηρόδρομο και στους αυτοκινητόδρομους, ενώ στα υπόλοιπα οι αυτοκινητόδρομοι λαμβάνουν ε, σημαντικό κομμάτι της χρηματοδότησης. Εάν δείτε όμως τους βασικούς στόχους του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής είναι ε, κατανοητό αυτό γιατί ο στόχος ε, είναι διαφορετικός στο, στο κάθε ταμείο και στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Όμως... Εάν συγκρίνεται τις δαπάνες με τους στόχους από το, τη Βίβλο για τις μεταφορές υπάρχει ένας κίνδυνος. Δηλαδή βλέπετε ότι όσον αφορά τις οδικές ε, μεταφορές φαίνεται ότι υπάρχει ένα είδος ε, στεγανοποίησης το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει τους περαιτέρω, περαιτέρω στόχους. Για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων υπάρχουν προτεραιότητες. Υπάρχει αυτή η επιλογή του 10% υψηλότερου δίκτυ συγχρηματοδότησης ανάλογα με τις διασυνοριακές ε, μεταφορές ή τους στόχους ως προς κλιματικές αλλαγές. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ως προς τις ε, διοικητικές ε, δυνατότητες υπάρχουν βασικές προκλήσεις να έχουμε με ένα σωστό ορισμό και προετοιμασία που δυστυχώς παρουσιάζουν αδυναμίες. Επίσης ήταν δύσκολο να ε, συνδυάσουμε το θέμα της διαδικασίας διαγωνισμών ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσα στα πλαίσια της συνέργειας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Και μιλάμε για αιρεσιμότητα εξ και έχει μεγάλη σημασία να δούμε κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα IPEC και JASPERS για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές ε, τις προκλήσεις καθώς και μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ του Jaspers και άλλων ε, ταμείων διαχείρισης. Στην ανάλυση που διενεργήσαμε βρήκαμε και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την ε, πολιτική στο σύνολό της, ίσως δηλαδή να μην αρκεί να θέσουμε μόνο μία σωστή πλαισίαση, θα πρέπει να υπάρξουν και άλλες προϋποθέσεις. Θα πρέπει να πληρούνται και άλλοι όροι. Δηλαδή, κατεξιοδότηση πράξης, οι, ε, τα, οι διάφορες κοινοπραξίες και συμπράξεις και ούτω καθεξής. Ως προς τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για την προτεραιότητα δαπανών στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Ταμείων, αν δούμε τους ε, στόχους μας, τους οικονομικούς και τους στόχους αντιμετώπισης των ε, κλιματικών αλλαγών, βλέπουμε ότι δεσπόζουν. Αν όμως δούμε πώς αποτιμούμε τις επιπτώσεις, βλέπουμε ότι στα σχέδια TEN-T το θέμα δεν είναι απόλυτα σαφές. Έχει μεγάλη σημασία να δούμε τι επιπτώσεις υπάρχουν και στον οικονομικό τομέα και στις κλιματικές αλλαγές. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε πιο αυστηρές προαπαιτήσεις, δηλαδή πρότυπα ε, συγκοινωνιών και μεταφορών, να αναλύσουμε και να αποτιμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές, ανάλυση κόστους ωφελίας, καθώς και ενιαία μεθοδολογία για την αποτίμηση του κόστους και της ωφέλειας. Αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί και έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς διενεργούνται όλα αυτά από ανεξάρτητους φορείς. Αυτά τα μέσα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την ιεράρχηση των σχεδίων. Ένα άλλο στοιχείο που μας απασχόλησε στην ανάλυση αυτή είναι η συνδεσιμότητα με άλλες πολιτικές έτσι ώστε να ορίσουμε τα διάφορα βάρη και τέλη, το ρόλο των υποδομών γιατί τα τέλη και οι επιβαρύνσεις μπορούν να διαδραματίσουν συγκεκριμένο ρόλο στη χρηματοδότηση των υποδομών. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε αυτά τα βάρη, αυτές τις επιβαρύνσεις. Αν δείτε όμως πώς αντιμετωπίζονται από το Ταμείο Συνοχής, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας αποτρεπτικός μηχανισμός ως προς την, ε, ως προς την ε, ε, τα, όπως προς τα βάρη αυτά κατά πόσο προσμετρούνται και ε, μπορούμε να πούμε ότι έμεσα τάσεται υπέρ των οδικών σχεδίων και κατά των σχεδίων για σιδηροδρομικές διασυνδέσεις. Όταν θέλουμε λοιπόν να συνδέσουμε τις διάφορες πολιτικές θα πρέπει να ορίσουμε προτεραιότητες. Υπάρχει λοιπόν συνδεσιμότητα μεταξύ ε, βαρών και τελών και ε, εξωτερικοποίησης του εσωτερικού κόστους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ αυτών των ε, πολιτικών, των στόχων. Υπάρχουν και τα, μέσα, τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης και η σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα για να δούμε ε, κατά πόσο και πόσο επιβαρύνεται ο δημόσιος τομέας. Επίσης θα πρέπει να δούμε ποιος ευεργετείται από αυτή τη δημοσιονομική πειθαρχία των ε, ιδιωτών επενδυτών έτσι ώστε να υπάρχει μία παγιοποίηση και οριοθέτηση καθώς και τυποποίηση των ε, μέσων καινοτόμου χρηματοδότησης. Πρόκειται για ένα περίπλοκο ζήτημα και νομίζουμε ότι δεν πρέπει να, προσθέσουμε όλα αυτά τα καινοτόμα στοιχεία, δηλαδή να τα δούμε σορευτικά. Τέλος, ως προς τα καινοτόμα μέσα, όπως τις ομολογίες για την χρηματοδότηση έργων, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να επιλύσουμε σε αυτή τη συνέργεια δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Τέλος, όταν δούμε την, το σύνολο των προτάσεων αυτών, θεωρούμε ότι έχει σημασία να ορίσουμε αυτό τον πυρήνα, το δίκτυο πυρήνα και παράλληλα Υπάρχουν κίνδυνοι που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ίσως βεβαίως θέματα χρηματοδότησης δεν έχουν επιληθεί πλήρως. Διανύουμε και μία περίοδο χρηματοοικονομικής ε, κρίσης που δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Γι' αυτό θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη και να δούμε ποια είναι και τα εναλλακτικά σενάρια, εάν υπάρχουν, για να δούμε τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Θα πρέπει να ορίσουμε ε, ένα κατά προτεραιότητα σχέδιο μέσα στα πλαίσια των ε, προσδιορισμένων εκ των προτέρων δικτύων, να δούμε δηλαδή με ποια, ποια είναι η βάση επιλογής αυτών των σχεδίων δηλαδή ε, ανάλυση κόστους ωφελίας, δείκτης ε, διοξιδίου του άνθρακα και ούτω καθεξής. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η εστίαση της προσοχής μας, της επιβαρύνσης επί του χρήση και τα εφή μέσα μεταφορών. Και βεβαίως να υπάρχει πλήρης αιτιολόγηση της ε, δαπάνης του δημόσιου χρήματος. Επίσης θα πρέπει οι επενδύσεις αυτές να υπηρετούν τους συγκεκριμένους στόχους, δηλαδή ε, λιγότερη έκκληση ιδιοξιδίου του άνθρακα και άλλη οικονομική στόχη. Αυτά εντάχει ως προς την μελέτη που διενεργήσαμε και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Βανέση. Έχουμε ένα κατάλογο 7 ομιλητών και έχουμε 25 λεπτά στη διάθεσή μας. 8 είναι οι ομιλητές μάλλον. Δύο λεπτά λοιπόν διαθέτεται ο καθένας προκειμένου να μιλήσετε όλοι. Ο κύριος Γκρός ε, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος Πρώτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες αυτές και θα ήθελα να περιοριστώ σε τρεις απλές ερωτήσεις. Πρώτον, περνάμε σε μια φάση πιλωτική των ομολόγων έργων που θα έχει αποφασιστική σημασία για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Δεν βλέπετε κάποια αντίφαση μεταξύ αφενός της προτεραιότητας, της ορίμανσης των έργων που συχνά βεβαίως εξαρτάται από τις δυνατότητες χρηματοδότησης και αφετέρου ε, στο διάφορους στόχους ε, είτε μιλάμε για κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή λοιπές πτυχές των μεταφορών. Δεύτερο ερώτημα Είχαμε και στο παρελθόν διάφορες ιδέες για τα οικονομικά μέσα. Θεωρείτε πως αυτά τα οποία προτείνονται όντως συμβιβάζονται με την οικονομική κατάσταση πολλών χωρών, όχι μόνο των γνωστών όπως της Ελλάδας, αλλά συνολικά με την κατάσταση. Έτσι ώστε ίσως αμφισβητείτε κάπως ε, η όλη αυτή η σύλληψη που μας παρουσιάστηκε τέλος ε, τα νέα μέσα, και εδώ πέρα βεβαίω εννοώ πάλι τα ομόλογα έργων, πώς τα βλέπετε σε σχέση με τα παλαιότερα. Ποια είναι η προσθέμενη αξία που προέκυψε από τη μελέτη σας. Είναι απάντηση στις αδυναμίες που διαπιστώσαμε στο παρελθόν ή είναι μόνο ένας νέος τρόπος έτσι ώστε να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμες ε, οικονομικές υποχρεώσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Αλχαντραβή για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Κάποια πράγματα. Είπατε πως είναι σαφές στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών το πώς θα συνεισφέρουν αυτά στην επίτευξη των στόχων της Λευκής Βίβλου. Από την άλλη, Αυτό δεν γίνεται, παραδείγματο χάρη, με τις τεχνικές ε, παρδιαγραφές, π.χ. για να είναι προϋπόθεση να συμμετέχει κανείς κάπου, να πάρει επιδοτήσεις από τα διευρωπαϊκά δίκτυα, το να έχει π.χ. περισσότερη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων και έτσι να έχουμε κέρδη ε, αποτελεσματικότητας. Το έχετε υπολογίσει αυτό. Έχετε κάνει κάποια μελέτη σε σχέση με αυτό. Βρίσκω ενδιαφέρον. Το ότι λέτε πως θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε άλλους στόχους ε, με κάποιες προδιαγραφές π.χ. όσον αφορά το εξωτερικό κόστος και την ενσωμάτωσή του. Ε, επίσης, ε, όπως ανέφερε και ο συνάδελφο, είμαστε σε δύσκολους ε, καιρούς δημοσιονομικού και μέσω άμεσης επιδότηση θα χρηματοδοτήσουμε μόνο ένα μικρό κομμάτι. Μπορούσαν λοιπόν να ληφθούν άλλα μέτρα τα οποία θα δυσκολεύουν τη δουλειά μας. Π.χ. σας δίνω ένα παράδειγμα, οι απαιτήσει κεφαλαιακές ε, όσον αφορά τα πιστοτικά ιδρύματα γίνονται αυστηρότερες. Τι αντίκτυπο θα μπορούσε αυτό να έχει σε, πρά... σε περιπτώσεις όπως τα ομόλογα έργαν. Τέλος, λέτε πράγματι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των στόχων ε, στους διάφορους μηχανισμούς στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα, έχουμε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κτλ. Μπορείτε να κάνετε κάποιες προτάσεις ε, σχετικά, κάποιες ιδέες για το πώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, μπορεί να εξαναγκαστεί να συνεργαστεί με, τον ίδιο τρόπο όπως ε, έχουμε εμείς κάποιους στόχους στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Να υπάρξει εκεί κάποια, να υπάρχουν κάποιοι όροι. Σας ευχαριστώ, Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση. Θα ήθελα να κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις. Βεβαίως είναι σαφές πως οι επενδύσεις οι οποίες ε, θεωρούνται απαραίτητες είναι προφανές πως δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν ε, από εμάς μόνο θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικού τρόπους χρηματοδότησης και βεβαίως ε, είναι και επιθυμητό αυτό Συγκεκριμένα θεωρείτε πως ε, με την καινοτόμο αυτή πρόταση έχουμε επαρκή κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα για να επενδύσει στα ευρωπαϊκά έργα. Και επίσης είναι σαφές πως ε, θα πρέπει να έχουμε κάποιους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Και το ερώτημα μου είναι θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποιοι άλλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης ε, τους οποίους δεν είχαμε σκεφτεί και θα μπορούσαν να είναι ενδιαφέροντες για τα έργα αυτά. Και βεβαίω. αυτό σχετίζεται με το ευρύτερο θέμα της δύσκολης οικονομικής κατάστασης και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ασχολείται με πολλές ρυθμίσεις του χρηματοοικονομικού τομέα. Σύντομα θα έχουμε και τη Βασιλεία 3, αλλά και άλλες ρυθμίσεις. Έχουμε την οδηγία περιφερειγκιότητας, στεξιοδοτικών ταμείων. Τι αποτέλεσμα θα έχουν όλα αυτά στη διαθεσιμότητα κεφαλαίου για αυτά τα έργα. Και τελευταίο, τελευταία ερωτήματα, μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας των ομολόγων έργου εξαρτάται βεβαίως ε, από την υψηλότερη αξιολόγηση, από τους οίκους αξιολόγησης και βεβαίως από τυχόν ε, δάνεια. Αν δεν γίνει αυτό υπάρχει ε, κάποιο plan B, κάποιο εναλλακτικό σχέδιο και τέλος ε, τα κόστος συναλλαγής και το διοικητικό κόστος το οποίο αναφέρατε στις ΣΔΙΤ δεν ξέρω αν θα υπάρχουν κάποιες ιδέες, κάποιες βέλτιστες πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στη συζήτηση. Φαντάλεν για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας. Θα αναφερθώ, θα κάνω κάποιες ερωτήσεις. Ε, όσον αφορά τα λεγόμενα αυτά ομόλογα έργων, μιλήσατε για κάποιο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα που θα έχουν και μιλήσατε για 15 πλασιασμό και 20 πλασιασμό. Πώς γίνεται αυτό ακριβώς, μπορείτε να μας εξηγήσετε. Πρώτον. Δεύτερον, για της ΣΔΙΤ, της Συμπράξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Ε, δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ μια, ένα πραγματικό πραγματικά επιτυχημένο ΣΔΙΤ ε, έχω ακούσει πάρα πολλά παράπονα. Μπορείτε να μας πείτε ε, αυτό είναι ένα υπόδειγμα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα. Και τέλος. στην εξέταση και τα συμπεράσματα της ε, πολιτικής. Ε, ίσως δεν σας κατάλαβα καλά. Βλέπω εδώ πέρα πως υπάρχουν δύο σκέψεις. Πρώτα μας λέτε πως ε, θα πρέπει να ε, υπάρχουν κάποια έργα προτεραιότητας, αλλά από την άλλη μας λέτε πως δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση. Ή παρανόησα, γιατί δεν μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό κάτι τέτοιο. Ε, αυτό το οποίο μας είπατε δηλαδή, για τα έργα προτεραιότητας και την ανεπαρκή χρηματοδότηση. Μάλιστα, ναι, ναι. Κύριος Κράμερ για δύο λεπτά. Εμείς συμφωνήσαμε πως η ενσωμάτωση του εξωτερικού κόστου θα πάει σε όλα τα μέσα μεταφοράς. Το ερευνήσατε. Εάν γίνει κάτι τέτοιο, πόσο θα κοστίσουν τα διάφορα έργα το εγκρίνομαι αυτό, μεγάλη πλειοψηφία, αλλά πρέπει να σημαίνει και κάτι να έχει συνέπειες για τη χρηματοδότηση. Δεύτερον, προσπαθήσατε τα νέα έργα ε, να οδηγήσουν σε κάποια αναβάθμιση κάποιων ε, ε δρομολόγιων. Να σας αναφέρω το σιδηροδρομο περολινο Βερολίνου-Αμβούργου που αναβαθμίστηκε και τώρα μπορεί να πιάσει το τρένο μία ταχύτητα 240 χιλιόμετρων την ώρα. Σε άλλα κομμάτια η ταχύτητα φτάνει 300 χιλιόμετρα. Αυτό συμπεριλαμβάνει, ε, ο υπολογισμός που έχετε κάνει συμπεριλαμβάνει το χρόνο και το χρόνο που γλιτώσαμε ή άλλα έργα που ολοκληρώθηκαν ε, πιο νωρίς. Τα έχετε υπολογίσει κατόπιν. Η έρευνα των διαδρομών και των διασυνοριακών διασυνδέσεων. Πόσα λεφτά έχουν πάει ακριβώς στα διασυνοριακά. Είναι πάνω από 3%, 5%, 1%. Πού έχουν πάει τα λεφτά στα εθνικά έργα, τα οποία κατ' ουσίαν είναι εθνικά και χρηματοδοτούνται ως ευρωπαϊκά. Εξ τώρα τα έργα τα οποία προτάθηκαν ε, με κάποια νούμερα, ε, τι έγινε τελικά στο τέλος και ανάλυση κόστος ωφέλους. Παραδείγματο χάρη υπάρχει σύγκριση των ε, οικονομικών, των οικολογικών συνεπειών π.χ. όσον αφορά το, το τούνελ στο Μπρένερ και την σύνδεση της Βαλτικής μήπως έτσι θα μπορούσαν κάποια έργα να είναι πιο πρώτης προτεραιότητας. Και τέλος, χρεώσεις, συγχρηματοδότηση μέσω των χρεώσεων. Λέτε, στον σιδηρόδρομο πρέπει κάθε τρένο να πληρώσει. Στους δρόμους, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ποια, ε, αν, είχαμε τέτοια τέλη θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Επίσης, για τις ε, ΣΔΙΤ, Ούτως ή άλλως ε, οι πιστώσεις ε, που δίνονται στον ε, ιδιωτικό τομέα είναι πολύ, με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από αυτέ οι οποίε δίνονται π.χ. στου Δήμου. Δεν το καταλαβαίνω γιατί. Κοιτάξτε, προσπαθώ να σφαιρίσω τα δύο λεπτά, αλλά βλέπω εδώ πέρα δεν με ακούει κανεί. Ο κύριο Κάντσιαν. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς, γιατί είμαστε σε μία στενοπό. Εάν τώρα ο καθένας ε, ε, τραβήξει προς τη δική του πλευρά, στην ουσία θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι δεν υπάρχουν δυνατότητες. Δηλαδή, ή χορηγούμε δάνεια με μία εγκυοδότηση ή κάνουμε επιδοτήσεις και συμμετέχουμε δωρεάν σε συγκεκριμένα σχέδια και προγράμματα. Αλλά τα ε, χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι τα ίδια. Γιατί όταν ε, μιλάμε για πολλαπλασιαστικό, ε, μάλλον για δίκτυ πολλαπλασιασμού, δεν θα πρέπει να θεωρήσετε ότι ξεκινάμε και φτάνουμε σε διαφορετικά ποσά. Δηλαδή, είτε γίνεται ε, δανειοδότηση και υπάρχει εγκυοδοσία, είτε δίνονται επιδοτήσεις. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο αυτά τα χρήματα έχουν δαπανηθεί κατά διαφορετικό τρόπο. Εάν θεωρείτε ότι για τις υποδομές μπορούμε να κινηθούμε με τους ίδιους πόρους, τότε Κάνετε μεγάλο λάθος. Εάν όμως η αγορά, στην περίπτωση αγοράς, αντί να στείλουμε τις επιχειρήσεις, στέλνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αλλάζει η ουσία των ομολογιών ε, δανεισμού. Γιατί σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ένα μηχανισμό εποπτείας σε αυτή τη δανειοδοσία. Και γι' αυτό, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να εκδοθούν ομολογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως. Αυτό εννοούμε όταν μιλάμε για project bonds. Η κυρία Τσικάου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Εντάχει, θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπονούντα τους εκπονούντες της μελέτης εάν λάβανε υπόψη την ε, διαμεσονομική εξυγίανση που ορίσανε τα κράτη-μέλη. Δηλαδή το γεγονός ότι ε, θα υπάρχουν επιπτώσεις σε δημόσιο επίπεδο των τεν τι. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω κάποια ερωτήματα για τους συντάκτες. Το βασικό μου ερώτημα είναι το γεγονός πως ε, στα μεγάλα έργα έχουμε κατά μέσο όρο 100%, 40 ε, με 100% υπέρβαση του κόστους. Ε, το ερώτημα λοιπόν είναι υπάρχουν εμπειρίες για το ποια είναι η επίδραση στη χρηματοδότηση γιατί είναι κρίσιμο ζήτημα. Γιατί σε τελική ανάλυση το κράτος μέλος ε, κάθεται με ένα σωρό απλήρωτους λογαριασμούς. Γιατί έχουμε πρόβλημα στο τέλος. Ή πληρώνουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια και το 40% της υπέρβασης που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχε γίνει καλύτερα η προκήρυξη του διαγωνισμού. Αυτό είναι βασικό για μένα. Δεύτερον, θεωρώ κάτι το οποίο είναι σημαντικό και στο ε, οι οικονομικές και κλιματικές επιπτώσεις δεν ε, έχουν υπολογιστεί σωστά στα περισσότερα έργα τα οποία υποβάλλονται. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα αξιοπιστίας. Πώς να πιστέψω παραδείγματο χάρη πως να πιστεψω παραδειγματος χαρη πως θα γίνουν παραδείγματος χάρη συνδέσεις πρόσβασης σε διάφορα διασυνοριακά περάσματα όταν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμα για τα τούνελ της ε, Ελβετίας ε, το οποίο ισχύει και για την Ιταλία και για τη Γερμανία αν δούμε τις Άλπεις. Τέλος, εγώ φοβάμαι λόγω αυτών των 10 δισεκατομμυρίων ε, για τα οποία πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης φοβούνται πως θα πάνε σε έργα στη Δυτική Ευρώπη ε, μπορείτε να αντικρούσετε κάτι τέτοιο ή όχι ή τέλος πάντων στο μεγαλύτερο μέρος θα πάνε τα 10 δισεκατομμύρια στη Δυτική Ευρώπη γιατί αυτοί είναι φόβοι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε γιατί πολλά από τα έργα τα οποία έχουν υποβληθεί είναι στα παλαιά κράτη-μέλη γιατί ε, βασίζονται στην παλαιά λίστα της ΕΣΥΣ. Οπότε το ερώτημά μου είναι υπάρχει η δυνατότητα να ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα. Τέλος, υπάρχει πρόβλημα στις λέξεις εδώ πέρα. Αυτή η υπόθεση με την καινοτόμο χρηματοδότηση Αυτό ε, κάπου αλλού, ξέρεις, ε, ξέρετε, έχει γίνει ταυτόσιμο της διαφθοράς. Λοιπόν, ο κύριος Κουμουτσάκος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συντάκτες της έρευνας. Είναι πραγματικά σημαντική. Δεν πάβει βέβαια να είναι σε μεγάλο βαθμό καταγραφική. Καταγράφει και αποτυπώνει μια κατάσταση όσο έχει. Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί το σύστημα χρηματοδότησης είναι πάρα πολύ σύνθετο. Και από εκεί πηγάζει η μία βασική μου ερώτηση. Ήθελα να ρωτήσω και για τα Project Bones, αλλά καλύφθηκα, καθώς και για τα Cohesion Funds, αλλά έχω καλυφθεί από προηγούμενους συναδέλφους. Λοιπόν, η βασική μου ερώτηση, γενική, προκύπτει ακριβώς από αυτή την μεγάλη πολυπλοκότητα του συστήματος χρηματοδότησης. Και σας ρωτώ σαφώς, εσείς πού εντοπίζετε τα προβλήματα και πού πιστεύετε και τι είδους διορθώσεις και βελτιώσεις μπορούν να γίνουν, ώστε και το σύστημα να γίνει απλούστερο, αλλά και ο συντονισμός αποδοτικότερος και μεγαλύτερος. Είναι μια σαφής ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μάισνερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται καν. Τρεις ερωτήσεις έχω. Εγώ νόμιζα πως ήταν 230 τα δισεκατομμύρια που θα ήταν τα ευρωπαϊκά κονδύλια ε, ε, από τα ομόλογα έργων για να προσελκύσουμε ιδιωτική χρηματοδότηση. Δεύτερον, για τα ομόλογα έργων μιλάμε για καινοτόμο χρηματοδότηση. Ε, βεβαίως από την άλλη λέμε πως υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα με την ε, ρευστότητα, τι θα μπορούσε να γίνει. Ποιος θα μπορούσε να μπει εδώ πέρα ως προς το χρηματοδότης. Και τρίτο ερώτημα, σωστά παρατηρήσατε πως ε, αυτή τη στιγμή πάρα πολλά έργα προτεραιότητας έχουν μείνει πίσω, εξού και η ρήτρα αυτή use it lose it. Το άμα τα αφήνεις αφήνει. Οπότε τι γίνεται, υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό όριο όσον αφορά την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία στο οποίο λέμε σε κάποια έργα δεν θα ισχύσει αυτή η αρχή ή πάει μετά όλο το έργο. Ο κύριος Ρικέ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι δεν θα μας φτάσουν τα χρήματα και ότι θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση. Πέντε ερωτήσεις έχω να κάνω σε σχέση με την διαιτησία. Πρώτον, ποια προτεραιότητα πρέπει να δοθεί ανάμεσα σε κάποια θέματα. Κεντρικό δίκτυο, παγκόσμιο δίκτυο, νέα έργα, εγκάρσια έργα, περιβάλλον, υποδομές. Δεύτερον, Είδαμε ότι το Ταμείο Φεντέρ είναι πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική χρηματοδοτική πηγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς μπορούμε λοιπόν να διαχωρίσουμε τρεις στόχους, σύγκληση, ανταγωνισμό και πώς θα γίνει αυτό όταν έχουμε κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται σε πολύ διαφορετικό επίπεδο ανταγωνισμού και τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε και με περιφερειακά ταμεία. Επίσης, τι απόφαση πρέπει να πάρουμε για την κατανομή των πόρων ανάμεσα σε ομόλογα, σε επιδοτήσεις και άλλα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Τέταρτη ερώτηση. Όταν ένα κράτο μέλος είναι επιλέξιμο όσον αφορά την, ένα στόχο σύγκλησης στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής καθώς επίσης και του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη, πώς μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στις τρεις δυνατότητες που πάντα υπάρχουν και τέλος για τα 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής, τα οποία θα δοθούν στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είναι κριτήρια του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη ή του Ταμείου Συνοχής ή θα γίνει μια επιλογή κριτηρίων και από τα δύο ταμεία. Και πώς λαμβάνεται υπόψη τις απαιτήσει που υπάρχουν στο κεντρικό δίκτυο, τις εθνικές απαιτήσει, καθώς επίσης και τις περιφερειακές ανάγκες και πώς γίνεται αυτό στα πλαίσια του Ταμείου Συνοχής, το οποίο παραμένει Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια του CEF. Ευχαριστούμε. Κύριε Βανέσε, θα ήθελα και εγώ να σας κάνω μία ερώτηση που έχει να κάνει με τη σύμπραξη δημοσίου τομέα. Όταν βλέπουμε τα ΣΔΙΤ σε πόσα από αυτά βλέπουμε τελικά να έχει ιδιωτικοποιηθεί το κέρδος και ποια από αυτά λαμβάνουν υπόψη και κάποιες κοινωνικές διαστάσεις. Έχετε το λόγο. Καλησπέρα. Ρόμπερτ Μπέιν ονομάζομαι κυρίες και κύριοι. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Ακούστηκαν πολλές, αλλά θα προσπαθήσω να συγκεράσω κάποια θέματα. Θα αναφερθώ στα ομόλογα έργων, στην σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα, στο ζήτημα των επιδοτήσεων και πώς μπορούμε να βγούμε από μια δύσκολη κατάσταση που έχει προκύψει. Όσον αφορά τα project bonds, τα ομόλογα έργων, ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό για μένα γιατί εργάστηκα στην Standard Reports για πολλά χρόνια και με ενδιαφέρει πάντα να δούμε ποιου βελτιωτικού μηχανισμούς μπορούμε να έχουμε για την δανειοδότηση. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα όσον αφορά, ε, δεν είναι ξεκάθαρα όσον αφορά την πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων. Καταλαβαίνουμε ποιο είναι ο βασικός στόχος. Να έχουμε δηλαδή ένα ομολογιακό δάνειο το οποίο θα προστατεύσει το βασικό τμήμα του δανείου, θα παρέχει κατά αυτόν τον τρόπο μία εγγύηση και κατά αυτόν τον τρόπο το senior debt θα μπορεί να έχει μία καλύτερη πιστολογική αξιολόγηση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ε, ένα κοινό έργο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από, για παράδειγμα, ιδιωτικά συνταξιδιωτικά ταμεία, από τον ιδιωτικό τομέα, από τις αγορές. Ξέρετε ότι υπάρχουν άλλοι οίκοι αξιολόγηση όπως η Moody's για παράδειγμα που δεν γνωρίζουν πολύ καλά τις λεπτομέρειες για τα project bonds και δεν είναι πεπισμένοι ότι θα δοθεί η βελτίωση δανειοδότησης ε, η οποία ε, θέλουμε να πετύχουμε μέσω των ομόλογων έργων και η Fitch ουσιαστικά έχει καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα ότι περιμένουν να δούνε τις ε, λεπτομέρειες και ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ακριβώς πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να σας πω και κάτι διαφορετικό όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις αγορές. Ένας από τους λόγους που έχουμε αυτή την πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργων είναι ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε τις απαραίτητες εγγύησεις μέσω των ασφαλιστικών οργανισμών που είχαμε στο παρελθόν. Και πολλές φορές ε, ξέρετε ότι προσπαθούσαμε να χρηματοδοτήσουμε διάφορα έργα μέσω ιδιωτικών συνταξιδοτικών ταμείων. Εκεί πέρα όμως ε, έπρεπε να υπήρχε μία πιστολογική αξιολόγηση. Βλέπουμε ότι πρόσφατα υπάρχουν από, τα, από το FSC ένα όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την χρηματοδότηση τέτοιων έργων και συνομίλησα με κάποιους επικεφαλείς από το FSC και μου είπαν ότι όντως θέλουν να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Επομένως υπάρχει πλέον η προοπτική να υπάρχουν ε, λιγότερες απαιτήσει για το όλο σχέδιο ομόλογαν έργων από ό,τι απαιτούσαμε στο παρελθόν. Κατά αυτόν τον τρόπο επίση μπορεί να γίνει μια αναβάθμιση τη αξιολόγηση για κάποια έργα και κατά αυτόν τον τρόπο διευκολύνονται οι επενδύσει. Η κατάσταση όμω είναι κάπω ασαφή αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα όσον αφορά τα ομόλογα έργων τώρα, όσον αφορά τη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Όσον αφορά τα ΣΔΙΤ λοιπόν, η ομάδα μελέτης είπε ότι είναι συγκρατημένα ενθουσιώδης σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή. Δηλαδή, είναι χρήσιμη αυτή η πρωτοβουλία εφόσον εφαρμοστεί σωστά και έχουμε κάποια παραδείγματα τα οποία δεν είναι θετικά. Γνωρίζουμε βέβαια ότι εμπλέκεται πάρα πολύ η πολιτική, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη σύγχυση, ενδεχομένως το ένα να πειράζει το άλλο, ότι υπάρχει και σημαντική έλλειψη ενημέρωση και πληροφοριών. Τα επόμενα δύο λεπτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε θα αναφερθώ ακριβώς στη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα και μπορούμε να το εξετάσουμε και την πλευρά της αξιολόγησης πιστολεπτικής ικανότητας αν δούμε ότι έχουμε δύο διαφορετικές εφαρμογές. Μπορούμε να δούμε τις οικονομικές υποδομές και τις κοινωνικές υποδομές. Και κάνω μια σαφή διάκριση με τις ε, οικονομικές ε, υποδομές, ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ πέρα είναι να δημιουργηθεί μεγαλύτερο κεφάλαιο. Δηλαδή, να έχουμε έναν μηχανισμό που θα μας επιτρέπει να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο κεφάλαιο και αυτό μπορεί να γίνει μέσω συγκεκριμένων έργων υποδομών, εισοδικέ μεταφορέ για παράδειγμα. Προσπαθούμε να βρούμε όμω κάποιε λύσει χρηματοδότηση αυτή τη στιγμή. Μέσω των τελών μπορούμε να έχουμε κάποιου νέου πόρου και αυτή η διάκριση μπορεί να γίνει ανάμεσα στην οικονομική και την κοινωνική υποδομή και τα ΣΔΙΤ χρησιμοποιούνται και για τα δύο. Στι κοινωνικέ υποδομέ δεν υπάρχει πληρωμή από του χρήστε. Επομένω εδώ πέρα έχουμε σχολεία, νοσοκομεία, έχουμε κοινωνική στέγαση, τέτοια προγράμματα. Πρόκειται λοιπόν για έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από δάνεια και για τα οποία απαιτείται μια χρηματοδότηση. Δεν δημιουργούνται δηλαδή νέοι πόροι ή νέα χρήματα. Προσπαθούμε ουσιαστικά εδώ πέρα να δούμε πώς μπορεί το κράτος να χρηματοδοτήσει τέτοια έργα για μια περίοδο 20-30 ετών. Έχουμε δηλαδή χρηματοδότηση από τον δημόσιο τομέα προς τον ιδιωτικό τομέα, προς τον φορέα παροχής. Σε πολλές χώρες υπάρχουν προβλήματα με αυτό το μοντέλο, για παράδειγμα στην ε, Πορτογαλία με τον ε, τομέα κατασκευής ε, αυτοκινητοδρόμων χρειάστηκε να γίνει μια μεταρρύθμιση όσον αφορά τη συμμετοχή του δημοσίου τομέα στον ιδιωτικό τομέα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων. Το σχέδιο αυτό δεν λειτουργούσε στο παρελθόν και είναι ακόμα πιο δύσκολο τώρα με την οικονομική κρίση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μάθαμε ότι θα βοηθηθούν κάποια σχέδια τα οποία στηρίζονταν στη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία νοσοκομείων. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα καταφέρουμε να εγγυηθούμε τις πληρωμές αυτές για τα επόμενα 20 χρόνια. Δεν υπάρχει όμως πολύ μεγάλη ευελιξία όσον αφορά την πολιτική που ακολουθείται για την συγκεκριμένη αυτή χρηματοδότηση, επειδή ακριβώς υπάρχει μια συγκεκριμένη δέσμευση πληρωμών. Και πολλές φορές οι οίκοι αξιολόγηση ακολουθούν πολύ, εκ του σύνεγγυς τι ακριβώς συμβαίνει σε ορισμένες χώρες, όπως για παράδειγμα σε κάποιες αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας, οι οποίες είναι όλο και περισσότερο εκτεθειμένες στις υποχρεώσεις που έρχονται στα πλαίσια συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Κάτι πολύ σημαντικό για μας είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα ΣΔΙΤ σας βοηθάνε να αγοράσετε πράγματα, όχι όμως να καταφέρετε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να καταβάλλετε τις απαραίτητες πληρωμές. και πώς μπορούμε τώρα να έχουμε τα απαραίτητα χρήματα προκειμένου να πληρώνουμε για τα σχέδια αυτά. Είτε πρόκειται για ΣΔΙΤ, είτε πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη μέθοδο χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ε, ένα συγκεκριμένος ρυθμός διαθέσιμων κεφαλαίων, τα οποία να μπορούσαν να δοθούν για μια περίοδο 20-25 ετών. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία προσπαθούν να βρουν τρόπους για να βαθμίσουν την υποδομή τους. Ακούνε πάρα πολλού οι οποίοι είναι οι θειασότε ε, των ΣΔΙ, των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα και εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε ότι δεν αποτελεί μία λύση μακροπρόθεσμη. Είναι μία λύση χρηματοδότηση που σα λέει απλώ πώ μπορείτε να αγοράσετε κάτι δεν σα εγγυάται όμω ότι θα έχετε σε ένα μεγάλο διάστημα χρόνου τα απαραίτητα χρήματα για να καταβάλει τι απαραίτητε πληρωμέ. Όσον αφορά τώρα τι επιδοτήσει, έχουμε εξετάσει το ζήτημα αυτό και στο παρελθόν και στα πλαίσια τη Επιτροπή Προπολογισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε κάποιε ε, πολύ ενθουσιώδει εξελίξει τα τελευταία πέντε χρόνια. Και αναφέρομαι εδώ πέρα στο loan grant blending ή τη συγχρηματοδότηση το συνδυασμό διαφόρων μεθόδων δανειονότησης. Αντί να παρέχεται απλώς μία επιδότηση, γιατί ξέρετε το πρόβλημα με την επιδότηση είναι ότι δίνεται χρήματα δωρεάν και αυτή είναι η αξία που τελικά δίνει ο κόσμος στο συγκεκριμένο έργο. Αν συνδυάσετε την επιδότηση αυτή με ένα δάνειο, τότε χρησιμοποιείτε όλους αυτούς τους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς προκειμένου να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση του έργου. Ας πούμε λοιπόν ότι τα Λάντερ έχουν μια επαγγελματική παρακολούθηση για το συγκεκριμένο αυτό έργο. Απαιτείται από αυτόν που έχει λάβει τα χρήματα να συμμορφωθεί, να πειθαρχήσει οικονομικά όσον αφορά την χρησιμοποίηση των χρημάτων αυτών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλυφθούν οι απαραίτητε διοικητικέ ευθύνε που συνδέονται με την αποπληρωμή των χρημάτων και το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε χώρε ή περιφερειακέ ή τοπικέ αρχέ στι οποίε δίνονται χρήματα συνεχώ χωρί να υπάρχουν κάποια κριτήρια χρησιμοποιώντας την μέθοδο αυτή συνδυασμού του δανείου με τις επιδοτήσεις, καταφέρνουμε να μειώσουμε το βαθμό της επιδότησης και να αυξήσουμε το βαθμό, το ποσοστό του δανείου με την πάρδο του χρόνου. Και κατά αυτόν τον τρόπο απεξαρτοποιούνται οι περιφέρειες, οι περιοχές αυτές από τις επιδοτήσεις. Διαφορετικά καταλήγεται σε μια κατάσταση όπου η επιδότηση διαιωνίζεται χωρίς συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία. Θα δώσω τώρα το λόγο στον συναδελφό μου. Yes, thank you very much. Also thank you very much for the, uh, uh, many and very... πολλά και ενδιαφέροντα ακούστηκαν. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα περισσότερα. Ελπίζω να μην ξεχάσω κάτι. Για το θέμα κατά πόσο υπάρχει αυτή η χρηματική δυνατότητα, μας ενδιαφέρει να δούμε τα, οικονομικά ωφέλη, τα ευεργετήματα ε, Αυτή της υποδομής. Γι' αυτό έχει σημασία να κάνουμε προβολές στον τομέα μεταφορών. Αν το δούμε αυτό στην Ολλανδία, πολλές φορές έχω την εντύπωση ότι ο έλεγχος συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι πολύ πιο δύσκολος και πολύπλοκος από ένα σχέδιο τεντή. Γι' αυτό νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Επίσης θα πρέπει να γίνεται μία ανεξάρτητη, ένας εξάρτητος έλεγχος ως προς, ως προς τη σχέση ε, ωφέλειας, κόστος ωφέλειας, προβολές ως προς τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες και ούτω καθεξής. γιατί υπάρχουν επιπτώσεις και στον ε, τομέα της έκκλησης άνθρακα. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες εκτιμήσεις και για τα δύο σκέλη. Αυτό είναι ένας απλός κανόνας που θα μπορούσε να προαπαιτείται. Δηλαδή, οι προαπαιτήσεις να είναι πιο συγκεκριμένες. Ως προς τα καινοτόμα μέσα, λέχθη μάλλον, μάλλον ρωτηθήκαμε κατά πόσο επαρκούν. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπορούν επαρκώς να χρηματοδοτήσουν, μπορούμε να δαπανίσουμε αυτά τα 540 δις. Μπορούν να δαπανηθούν σωστά. Δεν το ξέρουμε. Πάλι θα υπάρχουν θέματα χρηματοδότησης Γι' αυτό έχει σημασία να υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο, όπως είπαν και μερικοί. Πρέπει να υπάρχει ένα εναλλακτικό σχέδιο, εάν δεν μπορέσουμε, αν δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα ή εάν δεν αναπτύσσεται η οικονομία με τους ρυθμούς που πιστεύαμε μερικά χρόνια πριν. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα έτοιμο εναλλακτικό σχέδιο και να είμαστε σαφείς ως προς τις προτεραιότητες σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλήσαμε για το δίκτυο το οποίο είναι επικεφαλής και μετά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα εθνικά σχέδια με βάση αυτό τον πυρήνα, το δίκτυο πυρήνα. Αλλά δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα σε 10 χρόνια ή ίσως να μην μπορεί να γίνει. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει σωστή ιεράρχηση για το πώς κατανέμονται οι δαπάνες. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει περαιτέρω. Yes, I think this was covered already by you. Ως προς το, την ΕΤΕ, νομίζω ότι κάθε ταμείο έχει τις δικές του απαιτήσεις. Βεβαίως υπάρχει κάποια μορφή συνδέσμου ή σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις προτάσεις του TEN-T, διαρθρωτικά ταμεία του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα σημείο εκκίνησης και υπάρχει βεβαίως και σύνδεσμος με την ΕΤΕ σε σχέση με την ΕΤΕ. Είναι κάπως χιζοφρενικός αυτός ο οργανισμός. Θεωρείται ε, τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημόσιας ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αν δείτε τη συμπεριφορά της, ε, είναι μια επιθετική τράπεζα επενδύσεων. Εάν είναι τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε γιατί το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει την δυνατότητα να δει το πλήρες φάσμα δανειοδότησης της ΕΤΕ. Τα πρόσφατα χρόνια η ΕΤΕ δάνεισε ένα υπέρογκο ποσό, υπέρογκα ποσά, 70 δις ευρώ το 2010 μόνο. Θεωρείται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα είναι η μεγαλύτερη τράπεζα, αλλά η ΕΤΕ δανείζει 40% περισσότερο από την Παγκόσμια Τράπεζα σε ετήσια βάση. Όταν δούμε τα δελτία της ΕΤΕ, βλέπουμε ότι δεν ακολουθεί υγιή πολιτική δανειοδότησης. Πρόκειται για μια στοχοθέτηση, στοχοθέτηση ως προς τον όγκο του δανεισμού και τίποτα άλλο. Και ίσως θα πρέπει να σας απασχολήσει. Γιατί αν είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τότε εσείς θα πρέπει να την κατευθύνετε. Και εάν εσείς ορίσετε τις δανειοδοτήσεις της ΕΤΕ, τότε θα πρέπει να την απασχολήσει η ποιότητα δανειοδότησης και όχι τόσο η ποσότητα. Και εσείς να το κατευθύνετε αυτό. Ευχαριστώ, Ρόμπ. Ένα... Ένα άλλο θέμα αφορά τη δέσμευση των 10 δις και για το πώς αυτά τα ποσά θα δαπανηθούν. Θα δαπανηθούν και στη Δυτική Ευρώπη. Όχι αποτελεί μέρος της, όλα αυτά αποτελούν μέρος της, ε, του Ταμείου Συνοχής. Και υπάρχει η ίδια διαχείριση των 10 δις και του Ταμείου Συνοχής. Θα τα διαχειριστεί αυτά ο ίδιος ε, φορέας, ενώ για το Connecting Europe είναι ένα μέσο το οποίο είναι πιο ευρύ, ευρυδιαχείριστο. Ως προς τη διασυνοριακή διάσταση, τι δαπάνες θα γίνουν εκεί, καθίστατε σαφές στις νέες κατευθυντήριες γραμμές υπάρχει ένας κατάλογος προγραμμάτων και η κατανομή δαπανών. Δεν είναι απόλυτα σαφές, ε, υπάρχει ανταγωνισμός εκεί, αλλά οι κατευθυντήριες γραμμές και οι προτεραιότητες ως προς τη διασυνοριακή διάσταση είναι κάτι που, εντάξει, υπάρχει βέβαια, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, Όλα βρίσκονται επί χάρτου, αλλά πώς υλοποιούνται. Θα πρέπει τα χρήματα να δαπανούνται, να δαπανώνται κατά προτεραιότητα για αυτά τα σχέδια. Και οι συνολικοί στρατηγικοί στόχοι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά τώρα το τι γίνεται in situ, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο έγινε λόγος για ελέγχους εξ post, όμως θα πρέπει κυρίως να γίνονται εξ ante. Αυτά ίσως δεν απάντησα σε όλα, ελπίζω όμως τα περισσότερα. Ένα λεπτό, ένα λεπτό, Μάικλ. Μία ερώτηση είχα να κάνω όσον αφορά τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής, όσον αφορά τις προτεραιότητες, τα έργα προτεραιότητας που έχουν καθυστερήσει, καθώς επίσης και τη μη επαρκή χρηματοδότηση. Μάικλ, έχεις και εσύ μια συγκεκριμένη ερώτηση που δεν απαντήθηκε. Ναι, δεν απαντήθηκε. Για, τις... για την εμπειρία, μετά την εμπειρία με τα δύο συνοριακά κομμάτια. Τι ποσοστό ήταν. Ναι, τα ξέρω, ξέρω τους λόγους. Η ευρωπαϊκή υπεραξία είναι στο διασυνοριακό κομμάτι, αλλά δεν γίνεται. Και ποιο είναι το ποσοστό, αυτό είναι το ερώτημά μου. Αν ε, λέμε επίσης για εξυγχρονισμό εφιστάμενης γραμμής ε, και νέα κατασκευή. Ναι, μπορείτε να ξεκαθαρίσετε αυτό το θέμα και μετά βεβαίως και πού πάνε τα λεφτά. Αυτό είναι και σημαντικό ερώτημα. Μια στιγμούλα. ε, ναι, όλοι, όλοι το ίδιο θα πούν. Για το use it or lose it και την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, αν υπάρχει κάποια αντίφαση. Και αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Ναι, ναι, αυτό το τελευταίο ζήτημα δεν το κοιτάξαμε, η αλήθεια είναι πάρα πολύ λεπτομερός και δεν ε, υπάρχει και πολύ στην εκθεσή μας τους ήλους. Δεν μπορώ να είμαι λοιπόν πιο συγκεκριμένος. Θα το εξετάσουμε και ίσως μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάτι παραπάνω στην έκθεση. Για το δύο κομμάτι είναι σαφές πως στην τωρινή περίοδο χρηματοδότηση υπάρχει πρόβλημα με τα συνοριακά και ακριβώς αυτό είναι κάτι το οποίο τονίζουμε στην εξέταση της πολιτικής και και αυτό είναι ένας λόγος για τον οποίο ε, το λέμε συνέχεια. Πως πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα εκεί. Ένα από τα προβλήματα είναι πως καμιά φορά είναι δυσκολότερο να συντονιστούν αυτά τα δύο συνοριακά έργα. Οπότε το να λέμε μόνο ότι είναι προτεραιότητα δεν σημαίνει ότι γίνεται κιόλα. Είναι ένα πρώτο βήμα τουλάχιστον για να αποκτήσει μεγαλύτερη προτεραιότητα, υψηλότερη προτεραιότητα για το θέμα των ε, έργων προτεραιότητας που έχουν μείνει πίσω στο πρόγραμμα και της ανεπαρκούς χρηματοδότησης, αν συνδέεται αυτό. Ε, δεν ε, ξέρω αν ισχύει αυτό. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των δύο γεγονότων. Εγώ ήμουν και σύμβουλος σε κάποια έργα προτεραιότητας, ε, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης. Οπότε υπάρχει σαφής σχέση. Ε, χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί να, ξεκινήσει. Αυτή είναι η εξήγησή μου. Ελπίζω αυτή να ήταν η απάντηση που θέλατε να σας ικανοποιήσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω και στους δύο μιλητές μας, Βανέσεν και Μπέιν, ότι είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες που μας δώσανε. Πρόκειται για ένα σχέδιο μελέτης από το οποίο ακούσαμε. Δεν είναι η τελική εκδοχή της μελέτης. Προφανώς λοιπόν μπορούν να προσθεθούν και κάποια επιπλέον στοιχεία. Και ίσως και κάποια να πρέπει να αφαιρεθούν κιόλας. Πάντως είναι ενδιαφέρον ότι οι ευρωβουλευτές είχαν ε, πολλές ερωτήσεις. Ξέρω ότι η σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά πολύ. Ξέρω πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια PPP, Συμπραξιωτικού ιδιωτικού τομέα, που ουσιαστικά ιδιωτικοποιούν το κέρδος και κοινωνικοποιούν, αν θέλετε, το κίνδυνο. Πάντως είναι στη διάθεσή σας οι δύο μιλητές και μπορούν να σας δώσουν και περισσότερες λεπτομέρειες σε πιο συγκεκριμένε ερωτήσεις μπορεί να έχετε. Να σε ευχαριστήσω πάντως και τους δύο που ήρθατε εδώ και που μας εξηγήσατε αυτά τα πράγματα εγώ σίγουρα δεν έχω γνωρίσει κάποιον που να εργάζεται για αυτούς τους οίκους αξιολόγησης. Θυμάστε τους ε, οίκους αξιολόγησης που επικρίναμε στο Στρασβούργο πριν από δύο εβδομάδες, σας μην το ξεχνάμε. Πρώτη φορά λοιπόν για μένα. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπουμε στην ε, τελική εκδοχή της ε, μελέτης σας και προσβλέπουμε και σε μια μελλοντική επαφή μεταξύ ημών και των μελών της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Okay, so Antonio, you everything you need to Αντώνιο, τώρα ξέρεις τα πάντα όσον αφορά τα ομόλογα έργων. Και είναι ενδιαφέρον που ένας από τους κυρίους εδώ πέρα μας είπε ότι ο κύριος Μπένι συγκεκριμένα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να σου μιλήσει για τα project bond εφόσον το επιθυμείς. Το επόμενο σημείο είναι μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Προπολογισμών, συντάκτης γνωμοδότησης ο Αντώνιο Κανσιάν, γνωμοδότηση όσον αφορά τα ομόλογα έργων. Η Επιτροπή Προπολογισμών θα προχωρήσει πιο γρήγορα με την έκθεση αυτή. Ξέρω ότι δεν είναι α, όλες οι εκδοχές του κειμένου διαθέσιμες στα αγγλικά, πάντως πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί προχωράει γρήγορα και η Επιτροπή Προπολογισμών με το ζήτημα αυτό και Αντώνη σου δίνει ευθύς αμέσως το λόγο. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι θα χρειαζόμασταν περισσότερο χρόνο για ανταπαντήσεις, γιατί δεν είμαι ικανοποιημένος από τις απαντήσεις που έλαβα εγώ θα ήθελα να επιμείνω περισσότερο και νομίζω ότι η επίθεση κατά της ΕΤΕ θα έπρεπε να απαντηθεί. Πρόεδρος, τότε μέσω γραμματείας θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που μου είπε ο κύριος Μπέι είναι ότι αν θέλετε διασαφήσεις, εάν υπάρχουν ερωτήσεις, είναι στη διάθεσή σας να σας απαντήσει. Και έτσι θα έχετε την ευκαιρία να λάβετε μια απάντηση. Ωραία, ευχαριστώ. Σε σχέση με το θέμα μας που είναι συνέχεια των όσων ακούσαμε μέχρι τώρα, νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτή την ε, προτεραιότητα, με αυτή την πρωτοβουλία, με συγχωρείτε, των ε, project bonds. Γιατί Πιστεύουμε ότι είναι μια νέα πρωτοβουλία που αποτελεί διεύρυνση των LGTT που ήδη γνωρίζαμε που τροποποιούν τους κανονισμούς ε, του δημοσιονομικούς σε σχέση με το TEN-T και το TEN-N. Η ΕΤΕ εγγυάται την έκδοση ομολογιών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις των projects. Να το προσέξετε αυτό. Διότι πιστεύω ότι δεν προσαρμοζόμαστε σωστά στις συνθήκες. Πρόκειται Λοιπόν για εκδόσεις ομολογιών από τις ε, επιχειρήσεις των projects και έτσι ανοιχνεύεται καλύτερα το κεφάλαιο που χρειάζεται για τη χρηματοδότηση των υποδομών. Είναι ένα πολύ καλό πρώτο βήμα γιατί ανταποκρίνεται στις αγορές και στους εμπλεκόμενους φορείς που ενεπλάκησαν στις συζητήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα σχέδια τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν στην ιχνηλάτηση της σωστής οδού και του σωστού δρόμου που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Πρόκειται για ένα πιλωτικό σχέδιο που θα λήξει στο τέλος του 2013 μέχρι να αρχίσουν οι δημοσιονομικές προοπτικές 2014-20. Ε, έχουμε χάσει χρόνο, έχουμε χάσει ένα χρόνο και κάτι. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει η υλοποίηση το συντομότερο δυνατόν. Δεν λέω περισσότερα, διότι θα πρέπει καταρχήν να υπάρξει έγκριση Επίσης, ως προς τα 230 εκατομμύρια που έχουμε στη διάθεσή μας από το τέντι, νομίζω θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια διεύρυνση του πλαισίου, αλλά θα πρέπει να είμαστε και πιο φιλόδοξοι όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη που ελπίζω να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, εάν είμαστε ρεαλιστές δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα δίκτυα μεταφορών μόνο από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο στο CEF τα ποσά επαρκούν. Πιστεύω λοιπόν ότι οι ομολογίες έργων θα πρέπει να ισχύουν για μία βραχείο περίοδο και το business plan σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες θα πληρωθούν τη στιγμή που θα γίνει η εκχώρηση για τις υποδομές. Στην επόμενη παράγραφο όμως αναφέρεται κάτι άλλο. Τα περισσότερα σχέδια, για τα περισσότερα σχέδια όμως δεν καταβάλλονται τα χρήματα κατά τη στιγμή της εκχώρησης. Παλιά είχαμε μία άλλη δομή όπου στις περιφέρειες δίναμε grants, δίναμε επιδοτήσεις, αλλά τώρα έχουμε να κάνουμε με δημόσιο χρήμα. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση όπου θα πρέπει να προωθήσουμε τη δημόσια ανάπτυξη μέσω υποδομών. Για να βγούμε από αυτό το τούνελ. Κατά την άποψή μου λοιπόν αυτές οι ομολογίες έργου αποτελούν μια δημόσια έκδοση ομολογιών που από πλευράς επιχειρήσεων έργου δεν θα πρέπει εκεί να ε, δίνεται η ευθύνη, αλλά την ευθύνη τη φέρει ο δημόσιος τομέας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πρόκειται για χρήματα, για συγκεκριμένους στόχους υλοποίησης ευρωπαϊκών ε, διπονομών όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Δηλαδή, δεν πρόκειται για προτεραιότητες που μας επιβάλλουν άλλοι. Εάν λοιπόν υπάρχει σωστή διακυβέρνηση για την ε, υλοποίηση των έργων, όπως είπαμε χτες και για τα TEN-T, θα πρέπει εμείς ως Ευρωπαίοι συντονιστές να επιβάλλουμε προθεσμίες. Αυτό πέρα από τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Όμως η κάλυψη είναι αυτή. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τα χρήματα κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο και τελειώνουν κάποια στιγμή ή πάμε στην αγορά και αυτό μπορεί να γίνει χωρίς σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα, δηλαδή χωρίς το PPP. Πολλά χρήματα όμως λείπουν, γι' αυτό θα πρέπει να προσβλέπουμε στις αγορές. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Και έτσι ερμηνεύω την θέληση πολλών που θέλουν καινοτόμα μέσα. Αλλά αν δεν υπάρχει ε, χρηματοοικονομική βάση και πολιτική θέληση, δεν υπάρχει κανένα τεχνικό μέσο που θα, μας μπορέσει να, που θα μπορέσει να μας οδηγεί στην υλοποίηση αυτή. Η κυρία Γιάλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καντσάν και για τη μελέτη και για το νέο αυτό μέσο το οποίο ε, στην ουσία αποτελεί ε, πανεκκίνηση του LGTT. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μια, κατεπίγουσα, σε μια κατάσταση επίγουσας ανάγκης έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε ήδη, να αναγνωρίσουμε ήδη τους πρώτους επενδυτές. Θα ήθελα να υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις. Σε αυτή την πιλωτική φάση μπορούμε να προτρέξουμε κάπως και θα ήθελα να ξέρω για ποια projects μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι χρηματοδοτήσεις μόνο για τους διαδρόμους όπου υπάρχει χρηματοδότηση. Μόνο για το βασικό δίκτυο ή υπάρχει η δυνατότητα να επεκταθούμε. και στα συνολικά σχέδια και δίκτυα για να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν από πλευράς επενδυτών. Πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πύρα της ΕΤΕ σε σχέση με την προετοιμασία αυτών των σχεδίων που θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτών των χρηματοδοτικών μέσων και με βάση και τα μελλοντικά διευρωπαϊκά δίκτυα και μεταφορών και ενέργειας. Ποια, είναι η πείρα της ΕΤΕ και πώς μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα για τις χώρες συνοχής τη στιγμή που θέλουμε να διαθέσουμε άλλα δέκα δις από το Ταμείο Συνοχής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Θα μπορούσαμε επίσης να προετοιμάσουμε και τα σχέδια για την τρέχουσα χρηματοδότηση. Θα πρέπει όμως να ξέρουμε τι δυνατότητες υπάρχουν έτσι ώστε να είναι δελεαστικά αυτά τα σχέδια για μελλοντικούς επενδυτές. Ευχαριστώ και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Βεβαίω τα ομόλογα έργου είναι πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών μας γιατί βεβαίως δεν υπάρχει χρηματοδότηση από πλευράς ε, του δημοσίου και υπάρχουν και οι του προϋπολογισμού των κρατών. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε ιδιωτική χρηματοδότηση. Και θα πρέπει βεβαίως να υπάρξει και μια κάποια δημοσιονομική ε, πειθαρχία. Οπότε στηρίζουμε οπωσδήποτε αυτή την πρόταση και να ξεκινήσουμε αμέσως με τα πιλωτικά έργα και νομίζω πως και οι περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές θα είναι θετικοί, αλλά βεβαίως έχουμε κάποια ερωτήματα όσον αφορά τη διαφάνεια, την εφαρμογή όλων των στοιχείων των ομολόγων έργων και θα θέλαμε η Κομισιόν να κάνει μία αξιολόγηση για το πώς ε, μπορεί να είναι η εφαρμογή αυτών των ομολόγων, γιατί δεν επιτρέπεται να τρομάξουμε τους ε, ιδιώτες επενδυτές από το να επενδύσουν σε ευρωπαϊκές ε, υποδομές. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε, όπως είπα, το συντομότερο δυνατόν την πιλωτική φάση, αλλά με μία αξιολόγηση για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, καθισχάσουμε αποτελεσματικά τους ιδιώτες επενδυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Λίχτενμπεργκερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τα ομόλογα αυτά των έργων κατά τη δική μου άποψη και με βάση τα όσα ακούσαμε είναι ένα μέσο το οποίο δεν, ε, είναι, δεν ενδείκνυται για όλα τα έργα. Και το είπε ο εισηγητής. Όταν είναι πολύ μεγάλη διάρκεια, μέχρι πιθανώς να υπάρξουν κέρδη, το ερώτημα είναι ποιος πληρώνει και πού πάντα κέρδη. κατά το οποίο δεν είναι πάντα α, σαφές και δεν είναι πάντα ο ίδιος επίσης αυτός ο οποίος πληρώνει και αυτός ο οποίος ε, ε, καρπώνται τα κέρδη. Να δώσω παράδειγμα ε, επίσης όταν, κερδίζει, όταν γίνεται αυτοκινητόδρομο στο Τυρόλο δεν κερδίζουν οι ντόπιοι αλλά το Μόναχο με το Μιλάνο που συνδέονται καλύτερα και βεβαίως θα πρέπει να δούμε και την δυνατότητα που έχουν οι ιδιωτικοί όχι μόνο για την κατασκευή αλλά και για την εκμετάλλευση. Και εδώ πέρα ακριβώ είναι το πρόβλημα με το να υπάρχει δυσκολία στην εμπλοκή ιδιωτών επενδυτών γιατί θα πρέπει να υπάρχει μία ξεκάθαρη και άμεση παρουσίαση των, της σχέσης, αλλιώς δεν θα μπουν οι ιδιώτες επενδυτές. Αν μιλάμε για έργα τα οποία έχουν όντως μια πραγματική ευρωπαϊκή αξία, τότε έχουμε ακριβώς αυτό το ερώτημα. Γι' αυτό για μένα το θέμα αυτό με τα ευρωομόλογα ε, πραγματικά εξαρτάται από το να ορίσουμε ξεκαθαρά ποια είναι τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, ε, για να έχει νόημα. Και πρέπει να δούμε τι κίνητρα μπορούν να υπάρξουν και για το κράτος μέλος. Ε, π.χ. αν χρεώνεται η Αυστρία και μετά υποφελούνται οι δύο χώρες που ανέφερα, ε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και αν τα κέρδη μετά αναμένεται να φανούν σε 30 χρόνια, ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Αυτά είναι πράγματα. Να σκεφτούμε την πραγματική οικονομία που πρέπει να μας απασχολήσει. Αν σκεφτόμαστε μόνο τα κέρδη, εντάξει, είναι άλλο το ζήτημα. Μπορούμε να στείλουμε τα λεφτά βεβαίως να κάνουν κύκλους και θα κερδίσουν πολύ στο ενδιάμεσο. Αλλά εάν θέλουμε πραγματική χρήση στην πραγματική οικονομία, έχουμε δυσκολία εάν δεν ορίσουμε τους όρους ε, με μεγάλη ακρίβεια. Και αυτό το οποίο αναφέρθηκε και η σωστή χρηστή διοίκηση και η αξιοπιστία εδώ πέρα. Και είναι πράγματι ζήτημα αξιοπιστίας γιατί στην όλη αξιολόγηση χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουμε ζήσει αυτό. Γιατί? Γιατί μας τιμωρούν οι χρηματαγορές γιατί δεν είναι αξιόπιστο αυτό το οποίο προσφέρουμε. Ένα μέσο είναι βεβαίως η αξιολόγηση, αλλά πρέπει στο τέλος, στα συμπεράσματα να δούμε το μέγεθος, την ευκολία να μπουν οι ιδιώτες και πότε θα μπορέσουμε να έχουμε κέρδη, για να μην πάει όλη υπόθεση, στραβά. Και διεθνείς ε, επιχειρήσεις τώρα το να ενδιαφερθούν ενδιαφέρονται εκεί όπου υπάρχει κέρδος ποιος θα πληρώσει το κόστος και πόσο αξιόπιστη είναι η χρηματοδότηση. Και γι' αυτό έχω αμφιβολίες για το εάν εδώ θα καταλήξουμε κάπου. Δεν έχω δει εγώ ακόμα κάτι το έξυπνο και μια παρουσίαση σαφή των κριτηρίων από πλευράς κομισιών, γιατί αυτό το οποίο μου έχουν πει, κατά την άποψή μου, γιατί το είδα το, και το έδειξα σε ανθρώπους που ξέρουν από αυτά ε, και μου είπαν πως κανείς δεν θα έχει κίνητρο να εμπλακεί σε μια τέτοια υπόθεση. Μάλιστα. Κύριε Γκρός. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ε, κύριο Κάντσιαν έχω κάποιες τεχνικές ερωτήσεις. Τα κριτήρια επιλογής, αν κατάλαβα καλά, στην πιλωτική φάση είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται τώρα στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Ναι, όμως η συνεργασία ειδικά με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλάζει. Σημαίνει αυτό, μα, να το πω αλλιώς, εγώ δεν θα ήθελα να είμαι τόσο επικριτική όσο οι προλαλήσαντες ε, Ποιο είναι ακριβώς ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα είναι αποφασιστική η εμπειρογνωμοσύνη της για την επιλογή των τραπεζών ή τα υφιστάμενα κριτήρια είναι τα αποφασιστικά και μετά θα ε, πρέπει απλά να ελέγξει τη χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το πρώτο είναι αυτό δεύτερον. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια μέσα που πάνε παράλληλα και το LGTT ε, τι γίνεται, μπορούν να συνδυαστούν ή το ένα αποκλείει το άλλο. Το τρίτον, καλό είναι να μιλάμε για μόχλευση και για οικοσαπλασιασμό των κονδυλίων όπως ακούσαμε από την Κομισιόν. Δεν ξέρω αν σήμερα μπορούμε ακόμα να αναμένουμε κάτι τέτοιο. Και τέλος προς τον κύριο Κάντσιαν, στην έκθεσή του, εάν την κατάλαβα καλά, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα από τα ομόλογα έργου όσον αφορά την μείωση του κινδύνου αλλά και να περάσει κατευθείαν στη χρηματοδότηση των υποδομών. Θα με ενδιέφερε πώς, να δω πώς το βλέπει όσον αφορά την ευθύνη. Ποιος θα κάνει αυτό το βήμα και θα έχει την ευθύνη της χρηματοδότησης. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι εταιρείες που θα διευθύνουν αυτά τα έργα και οι ιδιώτες. Η κυρία Μάισνερ. Ja, danke schön. Also zum einen, ich denke mal, 2012, 2013 ist die Κοιτάξτε, 2012-2013 είναι η πιλωτική φάση, έχει ξεκινήσει, οπότε βιαζόμαστε λίγο για το εάν θα τα καταφέρουμε. Είναι φιλόδοξο αυτό το οποίο έχουμε, να δώσουμε 2,3 εκατομμύρια και να πάρουμε κάποια δισεκατομμύρια. Αυτό το οποίο είχε πει ο, Λιρέν. Οπότε απευθύνομαι απευθεία στην Κομισιόν. Αν είναι τόσο καλά τα πράγματα, μήπως να βγάλουμε περισσότερα. Γιατί θέλουμε να αποδείξουμε κάτι τέτοιο μέχρι το τέλος του 2013 και βεβαίω θα δούμε και τι θα υπάρχει μέσα στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Οπότε το ερώτημα είναι αυτά τα 32, τα 32 εκατομμύρια. Μήπως θα μπορούσαμε να δούμε ε, με τα λεφτά της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Τι, πρόκειται για μια μαγιά, εάν θέλετε, ε, μια σειρμαγιά για να μπορέσουμε μετά να προσελκύσουμε και τα κονδύλια των ιδιωτών αυτό είναι το νόημα, για να εξηγήσετε και τη λογική. Μάλιστα. Του απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον εισηγητή μας αναφερθώ σε ένα ζήτημα το οποίο αναφέρθηκε ο μιλητής μας ο κύριος Μπέιν στις απαντήσεις που έδωσε σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας. Αν αυτά τα ομόλογα έργων είναι κάτι το τόσο σημαντικό τελικά, για ποιο λόγο μέχρι στιγμής, μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι μας λένε ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και βλέπουμε ότι τα περισσότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι ιδιαίτερα διστακτικά και δεν θέλουν τόσο πολύ να δεσμευτούν. Ο κύριος Μπαρόζο είπε παλαιότερα ότι τα ομόλογα έργων ήταν η απόλυτη λύση για όλα. Και όταν συνεδρίασε η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, είδαμε ότι ουσιαστικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ένα συνδυασμό διαφορετικών συστημάτων. Ναι, τα project bond, αλλά και σε ένα βαθμό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τη σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Αλλά και εις δίτ πολλές φορές χρησιμοποιούνται υπερβολικά. Πολλές φορές ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιηθούν και λίγο πιο παραδοσιακοί τρόποι χρηματοδότησης έργων που αρχίζουν και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τώρα. Εγώ πάντως δεν θεωρούσα ποτέ, δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσαν τα ομόλογα έργα να αποτελήσουν μια θαυματουργή λύση για τα πάντα. Ποιος θα μιλήσει εξ ονόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Εσείς, ε, ποιος? Αποφασίστε ποιος από τους δύο θα μιλήσει. Μπορούμε να μιλήσουμε και οι δύο σύντομα. Συμφωνείς να, να αρχίσει ο μου και συνέχεια να συμπληρώσω κι εγώ. Ναι, πολύ ωραία. Ξέρω ότι είστε εμπειρογνώμονες στα πάντα, επομένως. Έχετε το λόγο. Σας ε, ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη που παίρνω εγώ πρώτος το λόγο. Ένα από τα ζητήματα που προέκυψαν από την παρουσίαση της μελέτης είναι ότι η εμπειρία με τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών δικτύων μέχρι στιγμής αποδεικνύει τελικά ότι υπάρχουν ε, διάφορα προβλήματα, διάφορες στενοποίοι όσον αφορά τη χρηματοδότηση, διοικητικά προβλήματα, έλλειψη συντονισμού. Αλλά είπαμε επίσης ότι δεν υπήρχε και η επαρκής χρηματοδότηση έργων. Αυτό τόνισε και η μελέτη. Πρέπει λοιπόν, προσπαθούμε με τα project bonds να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό μέσω των ομολόγων έργων. Προσπαθούμε να έχουμε επενδυτές ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία θα μπορούσαν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα μέσω των ομολόγων έργων. Προσπαθούμε λοιπόν να δεσμεύσουμε τα ιδρύματα αυτά, να χρηματοδοτήσουν τα έργα υποδομών, προκειμένου να αντικαταστήσουν ή να συμπληρώσουν την παραδοσιακή τραπεζική δανειοδότηση. Για ποιο λόγο λοιπόν οι τράπεζες αυτές οι οποίες μας δανειοδοτούσαν στο παρελθόν δεν μας παρέχουν το βαθμό δανειοδότησης που θα επιθυμούσαμε και στο μέλλον. Εν μέρει επειδή έχουμε την οικονομική κρίση και οι τράπεζες ήταν ο βασικός, η βασική πηγή χρηματοδότησης, δανειοδότησης στο παρελθόν έχουν αλλάξει πλέον συμπεριφορά πέντε στους νέους κινδύνους που έχουν, προ... που έχουν προκύψει και έχουμε και νέους ρυθμιστικούς κανονισμούς όσον αφορά τα κίνητρα για τις τράπεζες για να δώσουν τα απαραίτητα δάνεια. Νομίζω ότι πολλοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στα στοιχεία αυτά κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς ε, να συμπληρώσουμε κατά κάποιον τρόπο τη χρηματοδότηση αυτή, γιατί έχουμε σημαντικές φιλοδοξίες όσον αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών και θέλουμε σε ένα βαθμό να αντικαταστήσουμε την μειωμένη δανειοδότηση που προέρχεται πλέον από τις τράπεζες. Ένας ευρωβουλευτής πριν από λίγα λεπτά είπε ότι αυτή δεν είναι λύση για όλα τα έργα. Όντως, δεν πρόκειται για μία μοναδική λύση που θα ισχύσει για όλα τα έργα. Υπάρχουν πάντως ορισμένα έργα για τα οποία η χρηματοδότηση από τις κεφαλαγορές θα είναι δυνατή, ενώ για κάποια άλλα έργα δεν θα είναι δυνατή μια τέτοια χρηματοδότηση. Για τα έργα αυτά θα πρέπει να διατηρήσουμε τις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσει θα πρέπει να αποτελέσουν τον βασικό τρόπο χρηματοδότηση για κάποια έργα, ενώ θα προβλεφθούν παράλληλα και κάποιε άλλε μορφέ χρηματοδότηση. Υπάρχουν, όπω σα είπα, συγκεκριμένα έργα για τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και επιπλέον πόρους χρηματοδότηση, επιπλέον μεθόδους χρηματοδότηση. Ακριβώς στον τομέα αυτό λοιπόν προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα ομόλογα έργων. Και τα ομόλογα έργων δεν θα επιλύσουν όλα τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει όσον αφορά τη χρηματοδότηση υποδομών, όσον αφορά την ε, ε, λειτουργία της σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ούτε θα επιλύσει όλα τα προβλήματα που έχουμε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια πιλωτική φάση και χρησιμοποιούμε ως βασικό εταίρο την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν μπορούμε ουσιαστικά να βρούμε εύκολα εναλλακτικέ λύσει σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θεωρούμε πάντως ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτό φάνηκε και στη μελέχη, έχει δείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι είναι σε θέση να χρηματοδοτεί πάρα πολλά έργα. Όπως είπε και ένας ευρωβουλευτής, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει και να αναπτύξει τα έργα συνοδεύουν ουσιαστικά την υλοποίηση του έργου και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ένα συγκεκριμένο ισολογισμό μέσω του οποίου μπορεί να χρηματοδοτήσει την δική μας αρχική χρηματοδότηση. Μπορεί λοιπόν να αναλάβει ένα μέρος του κινδύνου και κατά αυτόν τον τρόπο είναι σε θέση η ΕΤΕ να προσελκύσει τους ιδιώτες επενδυτές. Ξέρετε ότι αυτοί οι ιδιώτες επενδυτές δεν προτίθενται αυτή τη στιγμή με ιδιαίτερο ενθουσιασμό να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση αυτών των έργων. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειε προκειμένου να του δελάσουμε, να του προσελκύσουμε. Και πολλέ φορέ, ακόμα και η καθυστέρηση που είχαμε στην υποβολή των προτάσεων αυτών οδήγησε στο να έχουμε ιδιώτε επενδυτέ, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα διστακτικοί και οδήγησε στο ότι υπάρχουν πολλοί και αξιολόγησεις οι οποίοι επιθυμούν στη φάση αυτή να εξετάσουν περισσότερο τι λεπτομέρειε. Εμείς θέλουμε όμως να καταφέρουμε να δελεάσουμε τα χρηματοπιστωτικά αυτά ιδρύματα, αλλά βέβαια θα πρέπει να εγκριθούν τα έργα, προκειμένου να μελετήσουν περισσότερο τις λεπτομέρειες. Αφορά λοιπόν συγκεκριμένα έργα και σαφώς η κατάσταση αυτή διαμορφώνεται έτσι εξαιτίας και της κρίσης και αποτελεί μια επιπρόσθετη μορφή χρηματοδότησης. Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη ε, πρόταση που έχει υποβάλει ο κύριος Κανσιάν, στην υφιστάμενη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, πρέπει ουσιαστικά να θέσουμε ένα ανώτατο όριο όσον αφορά την κεφαλαϊκή μας έκθεση. Ξέρετε ότι δημιουργούνται συγκεκριμένε ευθύνε μέσω του προγράμματο αυτού για τον κοινοτικό προπολογισμό. Ο κοινοτικό προπολογισμό δεν είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε να μπορεί να κρατήσει κάποιες μελλοντικέ ευθύνε, να μπορεί να συμπεριλάβει κάποιες μελλοντικέ ευθύνε. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ως μέσο του προπολογισμό και ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η ευθύνη που φέρει ο κοινοτικό προπολογισμό, θέτοντας ανώτατα όρια. η πρόταση αναφέρεται σε κάτι εντελώ διαφορετικό που θα πετούσε ουσιαστικά και μια επαναδιάρθρωση του κοινοτικού προπολογισμού ώστε να μπορεί να λάβει μελλοντικέ ευθύνε. Σε μια πιλωτική φάση δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όπω γνωρίζετε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τέτοιες Προσπαθούμε μέσω του κοινοτικού προπολογισμού να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα τη οικονομική ε, κρίση. Εγώ εξ ονόματος, για παράδειγμα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσπαθώ να εκδώσω ομόλογα και αυτό έκανε και στο παρελθόν για χώρες όπως η Ιρλανδία και δημιουργήσαμε συγκεκριμένες συνθήκες, εξαιρετικές συνθήκες ευθύνης για τον κοινωνικό προπολογισμό αλλά δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια διαχείρισης αυτών των ευθυνών. Δεν μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε σε αυτή τη φάση αυτόν τον δρόμο. Πρέπει να θέσουμε κάποια ανώτατα όρια και θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι η έκθεση, η κεφαλαϊκή έκθεση που έχουμε στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού. Διαφορετικά θα εκτεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σημαντικό οικονομικό κίνδυνο. Σα ευχαριστώ. Okay. Yes, thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ για να συμπληρώσω εντάχει για τα ίδια τα project, γιατί πολλά ανέκυψαν, δηλαδή ποια σχέδια θα, υποστηρίξουν αυτές, θα υποστηριχθούν από αυτές τις ομολογίες. Ε, πρόκειται για ένα μέσο από την εργαλειοθήκη που διαθέτουμε. Από την ε, προηγούμενη μελέτη που ακούσαμε νωρίτερα, βλέπουμε ότι ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι με τη συγχωρία των επιδοτήσεων με χρηματοοικονομικά μέσα. Γι' αυτό θα πρέπει σε αυτό τον αγωγό να ασχοληθούμε με τους πραγωγούς σχεδίων έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη όλο το φάσμα της εργαλειοθήκης όπως είπε και ο εισηγητής, για να βοηθήσουμε αυτά τα σχέδια, ώστε να είναι σε θέση να τύχουν χρηματοδότησης. Άρα στην ε, πιλωτική φάση τα σχέδια αυτά αφορούν όλο το φάσμα TNT, τα αρχικά σχέδια. Είναι σχέδια τα οποία καταρτίζονται ίδια, ήδη και η ασχολείται με τους προωθητές σχεδίων για να δούμε ποια σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτό που θα κάνει η Κομισιόν με την ΕΤΕ μέχρι το τέλος του έτους είναι να ασχοληθεί με μια στρατηγική προοπτική με βάση τις στρατηγικές προτερότητες του δικτύου που είναι ο πυρήνας και θα δούμε πού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το LGTT εκεί που χρειάζεται, τα project bonds και τις ε, επιδοτήσεις που προέρχονται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς ή από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TEN-T. Μιλάμε για την πιλωτική φάση, αν και είναι βραχύτατη φάση και θα πρέπει να συνεργαστούμε σωστά με την ΕΤΕ για να υπάρχει η σωστή ανάδραση από τη χρήση του μέσου αλλά ακόμα και αν δεν οριμάσει αυτή η διαδικασία στην πιλωτική φάση, τότε έχουμε το μέσο Connecting for Europe που πιστεύω ότι θα συνδεθεί επαρκώς, θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και θα μπορέσει να χρηματοδοτήσει αυτά τα καινοτόμα σχέδια. Μιλάμε για 200 ε, εκατομμύρια από το LGTT και πιστεύουμε ότι επαρκούν αυτά τα χρήματα για την πιλωτική φάση, για τα σχέδια και περισσότερα ποσά θα διατεθούν ε, από το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη κατά την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Ελπίζω να απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις και κάτι τελευταίο, για την διακυβέρνηση και τη λήψη αποφάσεων, αυτό το συζητήσαμε ήδη στην Επιτροπή και όπως είπαν και οι συνάδελφοι, μας ενδιαφέρει ο ισολογισμός του ΕΤΕ. Και εδώ έγκυται η ανάληψη κινδύνου. Γι' αυτό θα δούμε τι αναλαμβάνει η ΕΤΕ και θα δούμε κατά πόσο ε, αναλαμβάνει ένα μέρος της ευθύνης βεβαίως και η Επιτροπή και πιστεύω ότι μετά η τράπεζα θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε σχέση με την όλη διαδικασία πραγμάτωσης και υλοποίησης του project. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέσον. Τα θέματα χρονοδιαγράμματος είναι πολύ σημαντικά και χαίρομαι γιατί για, τα, ε, για τις ομολογίες έργων θα μπορέσουμε μέχρι το καλοκαίρι να αρχίσουμε με την πιλωτική φάση. Και μετά από την έγκριση, μετά το καλοκαίρι, θα ενημερώσετε την Επιτροπή για τα σχέδια που έχουν ληφθεί υπόψη στην πιλωτική αυτή φάση, για να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Καντσάν, θέλετε ε, κύριε Καντσάν, κάτι να πείτε εν συντομία. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσθέσω κάτι, γιατί η πρόθεσή μου δεν ήταν με αυτό το θέμα να διευρύνω το πλαίσιο και να πω ότι θα πρέπει να επεκταθούμε ε, προς την αγορά αλλά το σένσου θα έπρεπε να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο, αλλά και να αρχίσουμε μία συζήτηση για να δούμε κατά πόσο από πολιτικής πλευράς θέλουμε να στείλουμε στην αγορά αυτούς τους αναπτυξιακούς φορείς που προωθούν αυτά τα projects ή θέλουμε εμείς άμεσα να αποτανθούμε στην αγορά ως Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Αυτή είναι η επί της συζήτηση, γιατί φαίνεται ότι μπορούμε να πούμε ότι να δούμε, μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες ως προς τις υποδομές. Θέλουμε θεωρητικά, μιλάμε όμως για ομολογίες και στη συνέχεια την μεικτή το μεικτό αυτό φορέα να αποστέλουμε στην αγορά. Όταν μιλάμε για 200 λοιπόν εκατομμύρια που παίρνουμε από αυτό το σχέδιο δανειοδότησης του LGTT και τα παίρνουμε από εκεί τα χρήματα και λέω «Α, ένα μέρος το παίρνω από τα, τις ομολογίες έργου και ένα από το LGTT». Εάν όμως πάρω και από το μεν και από το δε, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αλλάζει το σύστημα χρηματοδότησης με βάση τα διαφορετικά μέσα χρηματοδότησης. Τι κάνω, προσελκύω ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτό που έχει σημασία είναι είτε χρησιμοποιήσουμε το ένα σύστημα είτε το άλλο, να δούμε ότι το σύνολο είναι αυτό. Υπάρχει θέληση λοιπόν για να πραγματοποιήσουμε ε, αυτή την ε, φάση εργασιών. Πώς γίνεται η χρηματοδότηση το 1993. Ο Ντελόρ μίλησε για δύο μέσα, δηλαδή ομολογίες της Ένωσης και μετατρέψιμες ομολογίες. Αυτά ήταν τα δύο μέσα. Μιλούσαμε ε, λοιπόν για ομολογίες μακροπρόθεσμες ομολογίες για την προώθηση στρατηγικών σχεδίων και οι άλλες ήταν μετατρέψιμες ομολογίες ε, σε μακρύ χρονικό ορίζοντα για να υλοποιηθεί το σχέδιο και που που την κάνουν εγγύησεις από κάποιο ευρωπαϊκό φορέα. Άρα τότε ο Ντελόρ είχε προβλέψει αυτές τις ομολογίες, τις μετατρέψιμες ομολογίες μέσα σε ένα μακροχρόνιο ορίζοντα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να μας απασχολήσει. Έχουμε να κάνουμε με ένα μέσο χρηματοδότησης εδώ, το οποίο προσελκύει κεφάλαια, αλλά σε ένα business plan που ε, λέμε ότι κινείται από 0 έως 100, θα πρέπει να δούμε μέχρι πού κινούμεθα για την εκχώρηση. Γίνεται η εκχώρηση, αλλά το υπόλοιπο του σχεδίου ποιος το χρηματοδοτεί. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει επαναφορά ή αντιστάθμιση όταν γίνει η επόμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος, δηλαδή ο επόμενος διαγωνισμός. Ευχαριστώ. Η προθεσμία είναι η 6η Μαρτίου και για τις τροπολογίες και στις 27 Μαρτίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα ψηφίσει Transport. στις 24. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καντσάν. Εμείς θα ψηφίσουμε στις 27 Μαρτίου. Τώρα προχωρούμε προς τους, με την ε, συνεδρίαση των συντονιστών. Διακόπτουμε για 10 λεπτά και στις 5 και 4 αρχίζουμε με τη συνεδρίαση συντονιστών. Σας ευχαριστώ.